Dear ladies, dear gentlemen, uh, thank you very much. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που είστε παρόντες στην ε, συνεδρίασή μας, η οποία μεταδίδεται και ζωντανά στο ίντερνετ και έχουμε διαθέσιμες 22 γλώσσες για διαρμηνία. Από χτες το πρωί δουλεύουμε μαζί με τους διαρμηνείς, Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε μια μισή ώρα τελειώνει όμως η συνεργασία μας. Θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Θα ξεκινήσουμε την κοινή μεικτή συνεδρίασή μας για το Mobile Health, την κινητή η υγεία, M-Health, είναι καυτό, καυτό θέμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι μεταδίδεται και στο ίντερνετ. Γιατί έτσι μπορούν να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις και οι πολίτες. Δύο ήταν οι βασικοί αίτη της μικτής αυτής, ε, της σύγκλησης της μικτής αυτής επιτροπής ο Αλόης Πέτρελε που εκπροσωπεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας, Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και ο κύριος Μπόνι που εκπροσωπεί την Ήτρα. Βιομηχανία, έρευνα, ενέργεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα όσα βλέπουμε δηλαδή στις ε, υπηρεσίες υγείας. μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες βεβαίως πρέπει να μεταχειριζόμαστε ως τμήμα της οικονομίας μας. Τούτων λεφτάντων, να δώσω το λόγο στον κύριο Πόνη, να πάρει τη θέση μου εδώ και εγώ θα πάρω τη δική του. Dear, dear colleagues, dear speakers. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι ο Τζοβάνι Λαβία. παρότι συμφωνώ με πολλές από τις ιδέες του και με μεγάλη μου χαρά εκπροσώπω την Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ουδέποτε είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω μία σύνοδο τέτοιες συνεργασίες μεταξύ των Επιτροπών Ήτρε και Ένβη με τον ε, ε, τέος ε, Πολωνό Πρωθυπουργό Γερζι Μπούζεκ σπάνιο να βλέπει κανείς δύο πρώην πρωθυπουργούς μαζί εδώ στη δουλειά αλλά έχω εδώ και την κύριο που θα πει πολύ σημαντικά μηνύματα αργότερα. Χαίρομαι λοιπόν που σας καλωσορίζω όλους εδώ στη σημερινή δημοσία ακρόαση με το θέμα της κινητής υγείας και το σχετικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Ειδικότερα θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και τους ομιλητές που θα μας δώσουν διάφορες οπτικές γωνίες για τις τεχνικές ε, πτυχές και τις πολιτικές πτυχές αυτού του πολύπλοκου θέματος και που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς θα επιτύχουμε κάποιους στόχους που σχετίζονται με την κινητή υγεία στην Ευρώπη από νομική άποψη, θεσμική άποψη. Θα μας μιλήσουν για τις απαιτήσει, διαλειτουργικότητες και τυποποίηση. Να πω ότι η κινητή υγεία δεν είναι ένα νέο πολιτικό σλόγγαν. Είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα καθήκον μια υποχρέωση και οι πολίτε το κατανοούν και καλωσορίζουν τις εξελίξεις προ αυτή την κατεύθυνση. Τα υγειονομικά συστήματα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν νέε προκλήσεις στη γύρανση του πληθυσμού και αυξημένη δημοσιονομική πίεση. Και σε αυτό το πλαίσιο η κινητή υγεία πιστεύω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Για πιο στοχευμένη ε, υγειονομική περίθαλψη, με εστίαση στην πρόληψη, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Και τώρα είναι τιμή μου και προνομιό μου να δίνω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Ανδρίου Κάιτης, αρμόδιο για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να μας ε, εκφωνήσει την ε, βασική την κυρία ομιλία του. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Πρόεδροι, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Και κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτό το εμπροστοβαρές γεγονό αυτή την εκδήλωση. Μιλάμε για κινητά πράγματα εδώ, όπως τα τηλεφωνά μας, με φαρμογές που είναι ιατρικής φύσης. Όλοι θα έχετε κάτι στα κινητά σας, δηλαδή θα έχετε την υγεία στην τσέπη σας. Οι ψυχακές τεχνολογίες και η γρήγορη ανάπτυξή τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την υγεία στην Ευρώπη. Οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και αποτελούν τμήμα της ψηφιακής επανάστασης. Οι ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται καθημερινά στη ζωή μας για την σωματική και ψυχική μας υγεία, την ιδιωτική και τη δημόσια παντού οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2013. Και σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς υπάρχουν πάνω από 165.000 εφαρμογές υγείας και ευημερίας από διάφορες πλατφόρμες. Αφορούν φυσική κατάσταση, τρόπο ζωής, αλλά και εφαρμογές με πιο περίπλοκες λειτουργίες που επικεντρώνονται σε ασθένειες και θεραπείες. Χρησιμοποιούν λοιπόν οι χρήστες των κινητών αυτές τις εφαρμογές στην καθημερινή του ζωή και αφορούν οι χρήσεις αυτές ε, κατανάλωση αλκοόλ, διαφορές δραστηριότητε, επιτείνουν διάφορες διαδικασίες και δραστηριότητε και βοηθούν και τις συλλογικότητες μέσω ας πούμε προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής. Και έχει βοηθήσει την αποτροπή ασθενειών υψηλό κινδύνου σε κάποιες κοινότητες αυτή η πραγματικότητα. Έχουμε μια εφαρμογή του iCoach που ήταν αντικείμενο της εκστρατείας μιας εκστατείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσε το κάπνισμα. Και 380.000 ε, καταγεγραμμένοι χρήστες ε, σταμάζαν το κάπνισμα μετά τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Έχουμε επίσης και θεραπείες με εφαρμογές που βοηθούν στην επίτευξη της θεραπείας και στην αποφυγή ιατρικών σφαλμάτων. Παρ' όλα αυτά, Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας βέβαια καμιά φορά για το κατά πόσο οι χρήστες είναι σε θέση να αποτιμήσουν τη χρήση τους και να κάνουν τις ε, κατάλληλες ενημερώσεις που θα τους βοηθούν στην υγεία τους. Θα πρέπει βεβαίως και αυτές οι εφαρμογές να συνδέονται με ιατρικούς φακέλους και να ενημερώνονται ιατρικά με την αυξανόμενη χρήση αυτό των εφαρμογών της χρόνιας παθήσεις και τη διαχείρισή τους θα πρέπει να μπορούμε να συνδέουμε τα δεδομένα με τους ιατρικούς φακέλους και αυτό αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά. Θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μικρά κενά. Θέλουμε να θεσπίσουμε έναν κώδικα διοντολογίας για αυτές τις κινητές, εφαρμογές κινητής και ε, τηλεφωνίας ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσει για τα προσωπικά δεδομένα. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση και ο κώδικας έχει μεταβαστεί στις αρχές προστασίας δεδομένων των χρόνο μελών. Θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω κατευθυντήριου για αυτές τις εφαρμογές, ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε διάφορα κριτήρια τα οποία θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία αυτών των εφαρμογών. Θα έχουμε προσεχώς ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για εφαρμογές υγείας. Αυτό θα το προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και Προτύπων. Επίσης θα έχουμε μια ευρωπαϊκή διαβούλευση για θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με τις εφαρμογές αυτές και επίσης για το λογισμικό για να ξέρουμε ακριβώς ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν γενικότερα στην χρήση αυτών των εφαρμογών και ειδικότερα στη χρήση των εφαρμογών υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τα επόμενα βήματα σε επίπεδο πολιτικών της Ένωσης. Οι χώρες μέλη αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών των διαφόρων δραστηριοτήτων και υπάρχει μια ομάδα εργασίας για την κινητή υγεία που σύντομα θα υποβάλει μια έκθεση για τις επερχόμενες προκλήσεις και τις πιθανότητες συνεργασίας μαζί με πρωτοβουλίες πολιτικής όσον αφορά χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας ώστε να προετοιμάσουμε σωστά και το επόμενο πρόγραμμα, πρόγραμμα 2000, ορίζοντας 2020 από το 18 μέχρι το 20. Να πω και δύο λόγια για την αυξανόμενη σημασία στα συστήματα υγείας αυτών των εφαρμογών και γενικότερα αυτών των εργαλείων και τι κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Είναι εργαλεία αυτά που βοηθούν τον εξυγχρονισμό των συστημάτων υγείας και τα βοηθούν να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις όπως γύραση του πληθυσμού και αύξηση των χρόνιων παθήσεων. Η ανακοίνωση του 2014 για προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας και η αντίστοιχη του 16 τονίζει το πώς ακριβώς μπορεί να ελοκληρωθεί η παροχή υγείας μέσω αυτών των εργαλείων ώστε να στοχεύουμε σε μια αποτελεσματική παροχή υγείας με την μείωση των σφαλμάτων και της νοσηλείας. Με την υλοποίηση λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων επικεντρώμαστε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε μικρή κλίμακα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές θα εφαρμοστούν όσον αφορά την διαδραστικότητα αυτών των εφαρμογών. Αν δεν υπάρχει διαδραστικότητα, σημαίνει ότι μια ηλεκτρονική συνταγή θα μπορέσει να μεταφερθεί διασυνοριακά. Και το ποσοστό νοσοκομείων που ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες είναι χαμηλό ιδιαίτερα διασυνοριακά. Και αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αυτά αποτελούν φραγμούς στην ελεύθερη, στην κυκλοφορία των ατόμων και οδηγούν σε κατακαιρματισμό της παροχής της υγείας του, της παροχής υγείας. Επίσης βέβαια έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της υγείας και πολλοί πολίτες θα πρέπει να σε θέση να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και να βοηθούνται από αυτά. Το 2015 είχαμε μια ανακοίνωση όπου ζητούσαμε περισσότερη διαδρασιμότητα και προτυποποίηση αυτών των εφαρμογών, διερευνώντας βεβαίως το, και αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό και τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές τις τεχνολογίες. Έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συνταγών και ιατρικών φακέλων ανά ασθενή διασυναριακά από 19 Απρίλη φέτος και μετά. Η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει μια υποδομή ψηφιακή η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη και υπάρχουν μεγάλες διαφορές βέβαια μεταξύ των χωρών μελών και αυτό ακριβώς η Κομισιόν προτίθεται να αναπτύξει, να, να υποβάλει έκθεση και συστάσεις. Η τηλεατρική είναι πολύ σημαντική εδώ στην χρήση αυτών των δικτύων. Τα δίκτυα αυτά έκπρος αντιπροσωπεύουν μια τελείως νέα προσέγγιση όσον αφορά τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Και η τελεατρική θα πρέπει βεβαίω να εφαρμοστεί δεόντως. Τα δίκτυα αυτά βεβαίως θα δημιουργήσουν και βάση δεδομένων για τους ασθενείς και να σας δείξω εδώ μια διαφάνεια Κόμπε, Ιαπωνία. Ο υπολογιστής Super K. Μια μόρφη υποδομής που δείχνει τη σημασία αυτών που συζητάμε. Η Ιαπωνία είναι έτοιμη ήδη να προχωρήσει και εγώ ονειρεύομαι, I have λέει ο μιλητής, να δω όλα αυτά να υλοποιούνται σε επίπεδο ένωσης. Ίσως να μην είναι εύκολο να συζητήσει κανείς όλα αυτά. Και ξέρετε τι δραστηριότητες έχουμε. Γαλιλαίο, Έρμπας και τα λοιπά. Είναι καλά παραδείγματα αυτά. Οπότε έχει έρθει η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και για αντίστοιχε υποδομές. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για έρευνα όσον αφορά τις ασθένειες, την αποτελεσματικότητα των θεραπείων κλπ. Επίσης εδώ θα έχουμε μια πρωτοβουλία που θα παρέχει στην ερευνητική κοινότητα μια παγκόσμιας κλάσης υποδομή για την αποθήκευση δεδομένων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παράσχουμε αυτή την υποδομή και για τα ιατρικά δεδομένα, οι δεδομένα υγείας, ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών. Καταλήγοντας, αυτά τα εργαλεία αποβλέπουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και θα επιτρέψουν στους πολίτες μας να βελτιώσουν την υγεία τους και να διαχειριστούν τις, την ίδια τους την υγεία. παραμένοντας πάντοτε βεβαίως συνδεδεμένοι στους παρόχους υγείας. Αυτά για το μέλλον. Και να σας πω ότι η Κομισιόν είναι τεθειμένη να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την κινητή υγεία το ταχύτερο δυνατό. Η κινητή υγεία λοιπόν αφορά το ερώτημα πώς θα προσεγγίσουν οι πολίτες την Ευρώπη. Η απάντησή μου είναι μέσω της υγείας φέροντας κοντά την Ευρώπη που αφορά την υγεία και την προστασία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε... Ευχαριστούμε πολύ για τα ξεκάθαρα μηνύματά σας Όπως είπα, οι πολίτες θα καταλάβουν τη δάσμευση που δείχνουμε όλοι, ώστε όλοι, όλες αυτές τις τεχνολογίες να είναι προσβάσιμες σε όλους και να τις χρησιμοποιούμε. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, αλλά οι συνεργάτες σας θα μείνουν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και καλή τύχη για αυτό το τμήμα, της, το επαναστατικό τμήμα της ψηφιακής ατζέντα. Επίτροπος, να πω και πάλι ότι ξέρετε έχουμε πολλά καλά project και πραγματικά παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και πολλών ε, μπλεκόμενων φορέων. Είναι λοιπόν σωστή η χρονική στιγμή να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτόν τον σούπερ υπολογιστή, τις υποδομές που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα, καινοτόμε θεραπείες, δυνατότητες να διαχειριστούμε την υγεία των πολιτών μας και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Έχουμε λοιπόν αξιότιμους προσκεκλημένους για να ξεκινήσουμε με, το, με την πρώτη σύνοδο και να δούμε τις ε, πιθανές, ε, τα πιθανά ωφέλη της ε, κινητής υγείας. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές μαζί μας σήμερα και θα δώσω το λόγο στον πρώτο, τον δόκτορα Άγγελο Κασιανό, μεταδιδακτορικό βοηθό ερευνητή στο UCL, για να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις για την υγεία στην Ευρώπη, για να θεραπεύσουμε και να, να προλάβουμε ασθένειες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε κιόλας σε μια πολύ σημαντική δημόσια κρόαση. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμες οι διαφάνειες. Πολύ ωραία. Θα σας δείξω εγώ την, ε, την οπτική του ερευνητή σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα που κάνουμε στο UCL. Θα σας ε, κάνω λοιπόν μια εισαγωγή. Αυτό μου ζητήθηκε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα στην υγεία και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την μετάβαση από την θεραπεία της ασθένειας στην πρόληψή της. Σίγουρα οι περισσότεροι γνωρίζετε τα στατιστικά στοιχεία. Είναι αυτά που δείχνουν ότι αυξάνεται ο πληθυσμός στην ε, Ευρώπη και αυτή είναι η βασική πρόκληση, τουλάχιστον σίγουρα μέχρι το 2020. Ε, ο γυράσκον πληθυσμό ε, έχει δημιουργήσει διάφορες προκλήσεις. Ζούμε πολύ περισσότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ζούμε υγιώς. Η υγιής ζωή μετράται από, τις, ε, από τα ποιοτικά προσαρμοσμένα ε, χρόνια ζωής. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορους ε, παράγοντες όπως χρόνιες ασθένειες, αλτσχάιμερ. Οι χρόνιες ασθένειες μάλιστα έχουν ένα 87% του μεριδίου των, της δημιουργίας προβλημάτων στη ζωή των πολιτών. Το κόστος όλων αυτών είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια οι περισσότερες από τις χρόνιες ασθένειες είναι ε, δυνατόν να προβλεφθούν. Να προληφθούν. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί ε, η κίνδυνη είναι ε, προβλέψιμη. Η, χρήση, η κατανόλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η ε, κακή διατροφή, η μία ε, άσκηση, εκείμναση Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε πιο εύκολα προσβάσιμα και πιο απλά συστήματα υγείας. Υπάρχει ε, μεγάλο προσδόκιμο ζωής με 10 ετών συγκεκριμένα για τις νέες χώρες. Μιλούμε λοιπόν για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες δημιουργούν μια δυνατότητα πολυεθνικής συνεργασίας και βεβαίως έχουμε, έχοντας υπόψη πάντα τα, ε, προ, τα ηθικά πρότυπα. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ είναι το άχθος των χρονίων ασθενειών. Ας πούμε για την Αφρική, όπου ο βασικός ε, ε, κίνδυνος ε, θανάτου είναι μεταδιδόμενες ασθένειες όπως η λονοσία και ο ιός του AIDS. Στην Ευρώπη είναι οι χρόνιες ασθένειες. Όταν μιλούμε για χρόνιες ασθένειες, μιλούμε κυρίως για ασθένειες όπως ο καρκίνος, η υπέρταση, ο διαβήτης, τα εγκεφαλικά κτλ. τα οποία ε, παίρνουν το 80% του μεριδίου του κόστους ε, στα συστήματα υγείας. Όλα αυτά βεβαίως είναι ε, δυνατόν να προληφθούν. Έχοντα λοιπόν υπόψη όλα αυτά και την έρευνα που γίνεται για την θεραπεία, έχουμε καταλήξει σε μία αλλαγή ε, και, επικεντρωνόμαστε πλέον στην πρόληψη της ασθένειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να πάει η χρηματοδότηση και στη θεραπεία των ασθενειών καθόλου. Σημαίνει ωστόσο ότι η πρόληψη των ασθενειών μπορεί να πάρει πλέον πιο πολύ προσοχή και να έχει και πιο μεγάλη χρηματοδότηση. Τι σημαίνει πρόληψη. Σημαίνει διάγνωση καταρχάς μιας ασθένειας, διάγνωση των συμπτωμάτων, των μηνυμάτων που μας δείχνουν ότι υπάρχει κάποια ασθένεια, έλεγχος του πληθυσμού και ε, τεχνικές ε, αλλαγής συμπεριφοράς των ασθενών. Ας πούμε, ε, αύξηση της άσκησης ή μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Και εδώ έρχεται το M-Health, η κινητή υγεία. Στην βιβλιογραφία λοιπόν το πιο χρήσιμο είναι οι απλοί ορισμοί. Αυτός ο ορισμός λέει ότι είναι οι πρακτικές υγείας κινητές και δημο... για τη δημόσια υγεία που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές. Ε, αυτό σημαίνει συλλογή δεδομένων για παράδειγμα. Τώρα προσπαθούμε να εκπονήσουμε μια εφαρμογή mobile health για να καλύπτουμε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα ζωής. Επίσης, παροχή ε, ε, πληροφοριών για την υγεία, ε, καλύτερη επικοινωνία ασθενούς και ιατρού, βοήθεια στους ασθενείς για να χρησιμοποιήσουν τα, τα φάρμακά τους, ας πούμε υπενθυμίσεις για να πάρουν τα, τα φάρμακά τους. Επίσης κλινικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι ιατροί που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εφαρμογές μέσω ας πούμε απάντησης ερωτηματολογίων. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ο αυτοέλεγχος του ασθενούς. Για παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ε, εκπονήσαμε μία ε, ε, εφαρμογή όπου ένας ασθενής μπορούσε να, πάρει, να βγάλει μια φωτογραφία ενός σπήλου για να ε, την δείξει στο γιατρό του και να δει ο γιατρός εάν αυτό μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να ε, ε, γίνει μελάνομα ή καρκίνος του δέρματος. Η PwC επίσης έχει κάνει μία έρευνα και αυτό που βλέπετε στις διαφάνειες είναι οι πιο συνήθεις απαντήσεις για το τι περιμένουν οι ασθενείς και ποιες είναι οι προτεραιότητες για την mHealth. Βεβαίως είναι το, κυρίως το πώς βρίσκω πληροφορίες, ε, πώς διαχειρίζομαι τις χρονικέ ασθένειες, πώς επικοινωνώ καλύτερα με τους παρόχους ε, ιατρικών υπηρεσιών, πώς διαχειρίζομαι την, ε, τα φάρμακά μου κτλ. Αν λοιπόν συνδυάσουμε όλη αυτή την έρευνα που όλο και περισσότερη είναι για την κινητή υγεία αλλά και τις συστηματικές αναθεωρήσεις και ελέγχους που γίνεται, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές συστάσεις στη βιβλιογραφία. Τα συστήματα λοιπόν M-Health πρέπει να ενταχθούν στα ήδη υπάρχοντα συστήματα υγείας διασυνοριακά. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται διαθέσιμα πρότυπα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ασθενούς. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχική προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κοινό, οι ασθενείς, οι ιατροί, θα πρέπει να εμπλακούν στη χρήση και στην, ε, καλύτερη, στον καλύτερο σχεδιασμό ίσως αυτών των ε, ε, εφαρμογών. Πρέπει να, είναι, υπάρχει ισοτιμία, πρέπει να είναι βιώσιμες αυτές οι εφαρμογές. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στην τεχνολογία, πρέπει να, να δούμε και τα αποτελέσματα και επίσης πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία, ας πούμε οι χαράζοντες πολιτικοί ε, εσείς για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορείτε να, κάνετε, ε, να πάρετε μια σωστή ε, εγνωσμένη απόφαση για αυτά τα θέματα σε ό,τι αφορά τη χάραξη πολιτικής. Και επίσης προσέθεσα κάτι που πρόσφατα είδα, γίνονται διάφορες μελέτες που λένε ότι πολλές ε, ότι οι εφαρμογές πρέπει να βασίζονται σε ε, φάρμακα που έχουν αποδείξει την ε, αξία τους. Πολλές φορές όμως αυτό δεν γίνεται και αυτό πρέπει να το προωθήσουμε. Τι σημαίνει τώρα αξιολόγηση του συστήματος ή του, της εφαρμογής mHealth. Σημαίνει, σημαίνει καταρχάς να αξιολογήσουμε δύο-τρία πολύ σημαντικά. Την ισχύ, δηλαδή κάνει αυτό που που προτίθεται να κάνει την αξιοπιστία, είναι αξιόπιστο σε διάφορα πλαίσια και περιβάλλοντα και είναι αποτελεσματικό. Πόσο αποτελεσματικό είναι τελικά στο τέλος. Έκανε όντως αυτό που έπρεπε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο δυναμικό να βελτιώσουμε τις, ε, την υγεία και τις ε, υπηρεσίες υγείας και κυρίως να, βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τον ασθενή. Την ποιότητα της ζωής τους για παράδειγμα μειώσουμε την, ε, τις, ε, τα προβλήματα, βελτιώνοντας τις διαγνώσεις ε, για τις χρόνιες ασθένειες. Βεβαίως υπάρχουν πολλές κλινικές δοκιμές που είναι πολύ εντατικές. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολλούς ασθενείς για να έχουμε πιο ασφαλή αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στην έρευνα, ένα μοντέλο προτύπων είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικά για να σας δείξω πόσο δύσκολο είναι και πόσο χρόνο και πόση χρηματοδότηση χρειάζεται για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα ότι κάτι, μια παρέμβαση, μια εφαρμογή mHealth όντως λειτουργεί. Για παράδειγμα, οι υψηλά, υψηλού επίπεδου ε, δοκιμές, έρευνα για την ε, διάδοση όλων αυτών των στοιχείων και κυρίως αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά το κόστος Ας πούμε, στα πλαίσια της εφαρμογής ε, αυτής της, ε, του application υπάρχει μείωση στο ε, τελικό κόστος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση που να πληρεί όλα τα κριτήρια αυτά. Δεν σημαίνει αυτές, ότι αυτές που υπάρχουν δεν είναι καλές, δεν είναι αξιόπιστες. Όχι. Αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αξιολόγηση αυτών των εφαρμογών, έτσι ώστε να έχουμε τελικά αποτελεσματικά συστήματα υγείας. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Αν ήθελα να σας δώσω ε, κάποια βασικά μηνύματα, θα ήταν καταρχάς να δημιουργήσουμε τη συνδημιουργία με τους ε, ιατρούς και το κοινό, να ε, μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε στην ε, στην δημιουργία τους. Επίσης ε, πολλές φορές υπάρχουν ιδέες αλλά δεν μένουν στο ράφι γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να ε, τις χρησιμοποιήσουμε. Επίσης πρέπει να έχουμε ασφαλή δεδομένα για να εκπονήσουμε τέτοιου είδους εφαρμογές και επίσης χρειάζεται υψηλού επίπεδου έρευνα για να Καταλήξουμε όμως αυτή την υψηλού επίπεδου έρευνα, χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι σε πολλές ε, σε πολλά, ε, σε, μεγάλη, σε πολλά τμήματα της νομοθεσίας για την ε, υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει έμφαση στην κινητή υγεία και βεβαίως πρέπει να υπάρξει μείωση των ανισοτήτων στην υγεία μέσω της mHealth. Ας πούμε, ομάδες που δύσκολα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους ασθενείς και το κοινό που δεν έχουν ας πούμε την οικονομική δυνατότητα να έχουν μια τέτοια εφαρμογή ή πιο ηλικιωμένοι. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισότητα στην ε, πρόσβαση στην, ε, στα συστήματα υγείας. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κασιανέ για την παρουσίασή σας. Με χαροποίησαν ιδιαίτερα τα μηνύματα κλειδιά και τα επισημαίνω και τα τέσσερα ότι η κινητή υγεία θα πρέπει να ελεγχιστοποιήσει τις ανισότητες στην υγεία. Εδώ στο Κοινοβούλιο είμαστε 751 ε, κλεγμένοι εκπρόσωποι των 500 εκατομμυρίων πολιτών ε, ε, της Ευρώπης και δεν τους αρέσουν οι ανισότητες, δεν τους αρέσει να τιμωρούνται αν δεν βρίσκουν γεννηθεί στο σωστό τόπο και ούτε μας μας αρέσουν αυτές οι μεγάλες διαφορές, αυτές οι ανισότητες. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι μια πραγματικά ψηφιακή προσέγγιση θα μας βοηθήσει να ελεγχιστοποιήσουμε τις ανισότητες αυτές με τη χρήση των νέων ευκαιριών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με χαρά μου τώρα να σας παρουσιάσω τον δεύτερο μιλητή τον Μάριο Μπορκόφσκι, ιατρό επικεφαλής ψηφιακής ιατρικής στην Adamet Group, θα μας μιλήσει για μια πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική ως προς το κόστος υγειονομική περίθαλψη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, το όνομα μου είναι Μάριος Μπορκόφσκι και προσωπώ εδώ την Adamet Group για να σας παρουσιάσω μια καινοτόμο μέθοδο για συντονισμένη υγειονομική περίθαλψη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πιστήσω στην προσοχή σας σε τρία γεγονότα. Το πρώτο, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, οι δημογραφικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε δραστικά υψηλότερες δαπάνες στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στο εγγύς Το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι ε, γινόμαστε όλο και πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία και πιο παγκοσμιοποιημένη. Το σημερινό σύστημα είναι κατακριματισμένο και οι ασθενείς ε, έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένες ε, λύσεις. Αναφέρθηκε και πριν λίγο εδώ μέσα στην αίθουσα. Το μέλλον θα απαιτήσει νέες λύσεις. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Αν προσθέσουμε στην υγειονομική περιθέλψη την σύγχρονη τεχνολογία, θα έχουμε προσθέμενη αξία και είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ναι, είμαστε έτοιμοι. σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ε, PwC και της σχετικής δοκιμής που ανακοινώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, το 60% των πολιτών της, ε, ε, των, χωρο, των κατοίκων της Ανατολικής Ευρώπης είναι έτοιμοι για την τηλεϊατρική. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της τηλεϊατρικής. Ναι, μια πλήρη μελέτη, η πιο πλήρης μελέτη, είναι η μελέτη Whole System Demonstrator του, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μελέτη αυτή βλέπουμε ότι ο σχετικός ε, κίνδυνος ε, εισαγωγής στο νοσοκομείο μειώνεται κατά 13% και ότι ο σχετικός κίνδυνος ε, θανάτου μειώνεται κατά 41%. Έχουμε και άλλη μια μελέτη από την Πολωνία που νομίζω θα είναι το πρώτο μέρος όπου ανακοινώθηκε τέτοια μελέτη και διεξήχθη από τον ε, καθηγητή Κριστάνεκ από το Πανεπιστήμιο της Ηλεσίας σε, με περίπου 290 ασθενείς ε, που υπέφεραν από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Η μελέτη διεξε 12 μήνες και ανέλησε όλες τις κλινικές παραμέτρους οι οποίε βελτιώθηκαν με τη χρήση τη τηλεϊατρική. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι το μέλλον θα απαιτήσει νέε λύσει. Θα χρειαστεί να συντονίσουμε την υγειονομική περίθαλψη και να προ... την εμπλουτίσουμε με την τηλεϊατρική. Υπάρχει κάποια λύση που θα μα βοηθήσει σε αυτό. κύριε και κύριοι, ναι, έχουμε λύση. Είναι το Μεντίβιο. Η Μεντίβιο, η πρώτη πιστοποιημένη κλινική τηλεϊατρικής. Δεν είναι άλλο ένα κατζετάκι από αυτά που βρίσκεται στην αγορά πολυάριθμα είναι μια πιστοποιημένη ιατρική συσκευή κατηγορίας 2α. Ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να θεραπεύσουμε ως γιατροί ασθενείς και το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, τις ε, ε, τηλεεπισκέψεις στο γιατρό. Όπως είπα, δεν είναι γκατζετάκι. Δεν είναι κάποια τηλεδιάσκεψη. Το Μεντίβιο είναι μια πιστοποιημένη ιατρική συσκευή, διαθέτει πιστοποίηση δηλαδή κλάσης 2α ως ιατρική συσκευή, ως ιατρικό μηχάνημα και έτσι οι ιατροί μπορεί να είναι βέβαιοι ότι η εξέταση, η διάγνωση και η θεραπεία που παρέχουν στους ασθενείς θα είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ιατρική περίθαλψη είναι η ανάκτηση των ιατρικών αρχείων διότι οι ασθενεί έχουν πρόσβαση ούτω ή άλλω σε αυτά τα ιατρικά του αρχεία, στο ιατρικό του ιστορικό, όποτε θέλουν και μπορούν να συμβουλευτούν αυτά τα δεδομένα μαζί με του γιατρού του διαφορετικών ιδιωτήτων, ειδικοτήτων, οι οποίοι χρειάζονται ενημέρωση, ε, και τι πληροφορίε αυτέ μπορούν να τι ανταλλάξουν ακόμη και μεταξύ χωρών. Έτσι, όπως είπα, μπορούμε να συλλέξουμε και δεδομένα και από τις κινητές μας εφαρμογές. Ε, σε όλους αρέσουν τα apps ε, και τα κατζετάκια, όλοι έχουμε. Οπότε από εκεί μπορούμε να συλλέξουμε τα δεδομένα αυτά. Για να συνοψίσω, τα χαρακτηριστικά του μεντίβιο είναι τέτοια που βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας θα επιστήσω την προσοχή σας ε, στα βασικά ωφέλη για τον ασθενή, για τον γιατρό και για το ιατρικό σύστημα. Για τον ασθενή έχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε ένα γιατρό μέσω τηλεεπίσκεψης ουσιαστικά. Για τον γιατρό το βασικό είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης το βασικό πλεονέκτημα είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία εφόσον χρησιμοποιείται το μεντίβιο, πιο αποτελεσματική θεραπεία με αποτέλεσμα οικονομία χρημάτων στο σύστημα υγειονομικής περιθάλψης. Ε, αποτελεί ενιαία πηγή επιδημιολογικών και στατιστικών δεδομένων, βοηθά στην παρακολούθηση τη ε, φαρμακοθεραπεία, υπάρχει ένα κεντρικό μητρό ιατρικών αρχείων online, υλοποίηση ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικών σημειωματών ασθενεία και ηλεκτρονικών παραπομπών και εισαγωγή τηλεεπισκέψη και τηλεδιάσκεψη. Ε, πράγματα που ανέφερε και ο κύριο Επίτροπο πριν από λίγα λεπτά. Τι γίνεται όμως με την ασφάλεια του συστήματος. Διότι μας απασχολούν φυσικά τα ζητήματα των ιατρικών στοιχείων. Είναι απολύτως ασφαλές, διότι όπως είπε ο συνομιλητής μου εδώ, είναι πολύ σημαντικό το σύστημα που θα χρησιμοποιούμε να είναι ασφαλές και το δικό μας σύστημα το μεντίβιο είναι ε, απολύτως ασφαλές. το αποδεικνύουμε αυτό με πιστοποίηση ISO και με την ε, κατηγοροποιήσει ω ιατρική συσκευή κατά κλάση 2α. Οπότε κυρίε και κύριοι, ένα όνειρο έχω. Το μεντίβιο να αποτελεί ε, αναπόσπαστο κομμάτι μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα τηλεϊατρική, όπου ο ασθενή θα βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο τη προσοχή. Το προϊόν αυτό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Αντάμεντ που είναι πρωτοπόρος ε, και καινοτόμος ε, της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Πολωνία και με τη Silver Media που είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία εργαλείων λογισμικού για τη διαχείριση ιατρικών διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι, από τη Μεντίβιο, την πλατφόρμα που επικεντρώνεται στον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Δεν είμαι ο μόνος που έμαθε κάτι νέο εδώ. Πολύ πιστικό και υποσχόμενο αυτό που παρουσιάσατε. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο για τρία λεπτά στη DG Συγγενική Διευθύνση Σάντε. Κύριε Αφίχα, από την Γενική Διευθύνση Σάντε και συνεργάτες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της ε, Κομισιόν. Α, ναι, αυτό ήταν το κουμπί, το βρήκα. Ναι. Είμαι επικεφαλής της ομάδας ηλεκτρονικής ε, υγείας και διασυνορικής υγείας. Όταν μιλάμε για υγεία διασυνοριακή, βασιζόμαστε σε μια οδηγία που όταν θα έχουμε εφαρμογές τηλεατρικής θα είναι όλο και πιο παρούσα στην πραγματικότητα. Αν έχουμε λοιπόν μια εξέταση τηλεατρικής διασυνοριακά. Αυτό μπορεί να αλλάξει τελείω τα πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι ακριβώ τονίζει το πώ τα δικαιώματα των ασθενών μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι εφαρμογέ αυτέ κινητή υγεία σα βοηθούν γιατί πραγματικά έχετε την υγεία στα χέρια σα. Αλλά νομίζω όταν, όταν αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται, η ηλεκτρονική και η κινητή, με τρόπο πιο κινητό, τότε οι ασθενείς έχουν περισσότερες δυνατότητες να ασχοληθούν με την υγεία τους, περισσότερο. Και για κάποιες χώρες του Βορρά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο οι νέοι ασθενείς δεν είναι αυτοί μόνο που αποφελούνται από αυτές τις εφαρμογές, αλλά όλοι οι ασθενείς. Αυτοί που συνήθω χρειάζονται περισσότερη περίθαλψη. Είδαμε κάποιες αποδείξεις αυτού του γεγονότος. Φυσικοθεραπεία, ας πούμε. Πώς θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω μηχανισμών, ίντερνετ δηλαδή, τηλεγιατρικής Ή ε, κι άλλοι, κι άλλες μέθοδοι μέσω εφαρμογών που βοηθούν ακριβώς την εφαρμογή της θεραπείας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση λέγοντας ότι η Γενική Διεθνή Υγεία συνεργάζεται στενά με οργανώσεις ασθενών. Θα έχουμε μια μεγάλη διάσκεψη σχετικά με την οδηγία συνολικής υγείας στις 24 του Οκτώβρη και εκεί ακριβώς θα παρουσιάσουμε κάποια πλεονεκτήματα που αυτές οι εφαρμογές κινητής υγείας έχουν για τους ασθενείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήσασταν πολύ καλός ευρωβουλευτής. Κατα, τα καταφέρατε ακριβώς το τρίλεπτο. Τώρα, λέει ο Πρόεδρος, πλησιάζουμε σαν πολύ σημαντικό κομμάτι της διάσκεψής μας δυνατότητα να σχολιάσουν. Έχουμε τον κύριο Κόκλησε, τον κύριο Σιλικιώτη από τους αδέλφους Βίρνιν και Κάλλας επίσης από την Άλντε. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Κόχλητσέκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ τους εισηγητές για τις παρουσιάσεις τους. Ε, στον κύριο Κόχλητσε έδωσα το λόγο πρώτα όμως. Ναι, δεν πειράζει παρακαλώ κυρία μου, συνεχίστε. Νομίζω, νομίζω ότι άκουσα το όνομά μου και παραξενήθηκα κιόλα. Τέλο πάντων, διαβάζω συχνά ότι πρέπει να υπάρχει διαδρασιμότητα μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών ακριβώς ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα. Τι γίνεται όμως με αυτή τη μεγάλη ποικιλία γλωσσών και ορολογία που έχουμε ανάλογα με την παθολογία. Θα πρέπει να μεταφράζονται αυτόματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο, κατά την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω κάποια πράγματα σε σχέση με το θέμα ασχολούμαι με καιρό, έχω γνωστού ε, γιατρού κλπ. Καταρχά να πω ότι η κοινή γλώσσα στην ιατρική είναι τα λατινικά. Αν υπάρχει συμφωνία για λατινική ορολογία δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά, στην Τσεχία προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε ένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υγεία. Αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο να ενοποιήσετε απλώς τους ιατρικούς φακέλους online, τότε και πάλι λύνεται το πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για λατινική ορολογία, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αγγλικά. Αλλά τα αγγλικά, ξέρετε, είναι και πολύ ευέλικτη γλώσσα. Κάθε λέξη έχει 20 ερμηνείε. Οπότε, ίσως θα πρέπει να βρούμε μια άλλη γλώσσα. Ίσως, ας πούμε, πολύ ακριβής γερμανική γλώσσα. Θα ξαναπώ λοιπόν ότι η βάση για την ανταλλαγή δεδομένων είναι ένα κοινό πρωτόκολλο. Όπως συμβαίνει παντού στην τεχνολογία των υπολογιστών. Θα πρέπει βέβαια να καθορίσουμε τι σημαίνει τι, λατινικά οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Επίσης, να πω ότι αν συμφωνήσουμε τελικά, ας το κάνουμε αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να έχει το δικό του φάκελο μαζί του, διαθέσιμο γιατί βεβαίως και οι σερβερ δέχονται επιθέσεις και τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται με ένα ενοποιημένο πρωτόκολλο μπορούν να δεχτούν ηλεκτρονική επίθεση, έτσι. Θα ήταν λοιπόν καλό κάθε ασθενής να έχει το δικό του φάκελο μαζί του. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και ο Πρόεδρος. Κάποιος άλλος μήπως. Από την κοινωνία των πολιτών, πού είσαστε, εδώ είσαστε. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Αναρωτιόμουν. Όλα αυτά περιλαμβάνουν και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό σκοπό, όπως δείξατε. Συχνά το συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο Υπάρχει μια αντίρρηση γι' αυτό. Ότι φοβάται ο κόσμος κατάχρηση των δεδομένων τους και τα δεδομένα υγείας είναι τα πιο ευαίσθητα. Είναι όμως και δεδομένα τα οποία βοηθούν περισσότερα απ' όλα. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή την διαφορά, αυτή την αντινομία, δηλαδή κάποιος άλλος να μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά ιατρικά δεδομένα Ευχαριστώ πολύ. Μήπως κάποιος από το πάνω θα ήθελε να απαντήσει. Ο κύριος Κασιανός. Ναι, αυτό πραγματικά είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε συνεχώς στην έρευνα. Η διαχείριση των δεδομένων όχι μόνο για τα μεγάλα δεδομένα σε αυτό το πεδίο και δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση, αλλά θα έλεγα για να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προς τους ασθενείς και το κοινό για το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ας πούμε, άμα θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πρωτόκολλο Διοντολογία που λέει ότι ποιος θα χρησιμοποιεί, ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα, πώς τα δεδομένα μετά θα κυκλοφορήσουν. Από τη δικιά μας ερευνητική εμπειρία αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή, από τους χρήστες αυτών των δεδομένων, από τις πηγές αυτών των δεδομένων. Δηλαδή ποιος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τους. Αλλά συμφωνώ, δεν είναι απλό το πρόβλημα, είναι θέμα αρκετά περίπλοκο και νομίζω ότι έχει να κάνει με διάφορους κανονισμούς και διάφορες προσεγγίσεις στις χώρες σε σχέση με την αποθήκευση δεδομένων ή την χρήση τους. Υπάρχουν όμοι τρόποι παράκαμψης του προβλήματος και ένας από αυτούς τρόπους είναι το να καταστήσει σαφές από την αρχή το τι κάνεις. Ναι, και εμείς για το προϊόν μας ενημερώνουμε με διαφάνεια τους ασθενείς ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από σερβερ. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα συστήματα. Είναι ανώνυμα αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιούνται σε κάποια ιατρικά προγράμματα και παροχής υπηρεσιών υγείας χαρτογραφώντας δηλαδή τις ανάγκες των ασθενών, βοηθώντας τον πληθυσμό μακροπρόθεσμα. Νομίζω το πιο σημαντικό εδώ είναι να είναι κανείς διαφανής, και να προκαταβάλει ακριβώς τον τρόπο χρησιμοποίηση των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ και Πρόεδρος. Στο Μιχαλ Μπόνι, το συνάδελφο, θα δώσω τώρα την Προεδρία, ο οποίος θα παρουσιάσει το επόμενο σημείο την επόμενη συνεδρία. Τη δεύτερη. Η σειρά σου είναι. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε στον περίνα του ζητήματος εδώ γιατί η δεύτερη αυτή συνεδρία λέγεται ξεπερνώντας τους φραγμούς την εφαρμογή της κινητής υγείας τα δεδομένων, διαλειτουργικότητα. Να καλέσω τον κύριο Άιν Άβιξον, αναπληρωματικό, αναπληρωτή γενικό γραμματέα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την καινοτομία από το Εσθονικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και τον κύριο Μικέλε Παστόρε από το Digital Europe ε, και την Ομάδα για την Ελεκτρονική Υγεία. Βρισκόμαστε εδώ σε μια φάση εφαρμογής, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν 54 επιλογές για τις χώρες μέλη όσον αφορά την εφαρμογή. Αυτό αφορά και το τομέα της υγείας, όπου χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση. Ας πούμε, φοβόμαστε ότι κάποιες χώρες θα επιλέξουν διαφορετικό δρόμο από άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι που στο Κοινοβούλιο και στη συνεργασία με τις Εθνικές ε, Βουλές θα πρέπει το 17 να πείσουμε τους αδέλφους ότι θα πρέπει να έχουμε κοινέ λύσεις. Εντάξει, υπάρχουν κανόνες για ανωνυμία ή ψευδονυμία των δεδομένων. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συζητηθεί εδώ στην συνεδρία μας. Να δώσω καταρχάς το λόγο λοιπόν στον κύριο Άιν Αά ο οποίος θα μας μιλήσει για την προστασία των δεδομένων, ιδιοκτησία και φορητότητα. Και για ένα νέο κώδικα διοντολογία για αυτές τις εφαρμογές κινητής υγεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, με χαρά και τιμή είμαι εδώ και όταν είδα αν δείτε μάλλον τον τίτλο της παρέμβασής μου είναι μακρύς αλλά το μήνυμα είναι βραχή. Ναι, ξέρουμε και έχουμε πλαίσια αλλά θέλουμε να δούμε αν είναι σωστά. Να σας δώσω κάποιες κατευθυντικές γραμμές γενικά. Πρώτα, ακούσαμε ήδη ότι η περίθαλψη αλλάζει. Έχουμε συστήματα υγείας ακόμα όπου ακολουθούν μια πυραμίδα όπου έχουμε κυρίως τα νοσοκομεία με τεχνολογία και την περιθάψη των πολιτών, οι οποίοι βεβαίω εύχονται ότι εκεί θα θεραπευτούν. Τώρα βέβαια έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις ανά σύστημα υγείας. και υπάρχουν όλο και περισσότερο υπηρεσίες, υπηρεσίες βοηθητικές και που βοηθούν στους ασθενείς στο σπίτι και χρειάζονται αυτά τα δεδομένα και αυτά τα εργαλεία που αναπτύσσουμε. Τώρα θα πρέπει να αναζητήσουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση δηλαδή κόστους ωφέλους, να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία και αποδείξεις και όλα αυτά σε με μια εξατομίκευση αυτών των παροχών. Δηλαδή όσον αφορά τη διαχείριση από κάτω προς τα πάνω της υγείας και τις παροχές μονάδων υγείας προς τους πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουμε και ακριβώς την πιο αποτελεσματική μορφή υπηρεσίας υγείας ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Ήδη ακούσαμε ότι εδώ η καινοτομία και μία από τις προηγούμενες εισηγήσεις το ανέφερε αλλά να σας πω ότι και η Κομισιό Χρηματοδοτή αντίστοιχα προγράμματα και οι χώρες θα πρέπει βέβαια να το χρησιμοποιήσουν αυτό, γιατί αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Να σας πω λοιπόν ότι δεν ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζω να διαβάσατε κάποια από εσά την έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από 4,5 χρόνια από την ομάδα εργασία για την ηλεκτρονική υγεία. Ο κύριος Αλκίδης ε, προέδρευσε σε αυτή την ομάδα. Παρατήθηκε πριν από λίγες μέρες και πήγε στην Εστονία. Στη μελέτη αυτή προσπαθήσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπους ώστε η υγεία να είναι λιγότερο παρεμβατική και πιο αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος. Και τι βρήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν ότι καταρχάς η υγεία είναι κάτι πολύ προσωπικό για να κάνουμε λοιπόν τις πληροφορίες και τα δεδομένα χρήσιμα για τους ανθρώπους και την υγεία τους, θα πρέπει αυτοί να έχουν τον έλεγχο αυτών των δεδομένων. Οι αποφάσεις των ασθενών και τα αντίστοιχα δεδομένα θα πρέπει να διευκολύνονται σε συνεργασία, σωστή συνεργασία με τους επαγγελματίε της υγείας, αλλά και με ειδικού, που δεν σημαίνει απαραίτητα γιατρούς και νοσοκόμες. Δεύτερον, είδαμε επίση ότι σε αυτή την πυραμίδα που είδαμε προηγουμένως στη διαφάνεια, τα περισσότερα δεδομένα παραμένουν σε αυτού του θεσμού, Δεν μετακινούνται και αυτό για διάφορους λόγους. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή τα δεδομένα θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των διαφορών θεσμών και όπως ακούσαμε διασυνοριακά μεταξύ κρατών. Τρίτον, είδαμε ότι αυτά τα συστήματα ολοκλήρωσης που είναι διαφορετικά από την πυραμίδα μπορούν μόνο να λάβουν χώρα μόνο αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προωθήσουμε με την συνδεσιμότητα μέσω κινητού ή μέσω τηλεκοντρόλ ή τηλεελέγχου αυτών των δεδομένων, ώστε τα δεδομένα αυτά να είναι ενσωματωμένα στο σύστημα. Ακούσαμε επίσης ότι έχει έρθει η ώρα, υπάρχει η τεχνολογία, έχουμε καλά παραδείγματα από άλλα μέρη του κόσμου, οπότε απλά και μόνο χρειάζεται να κάνουμε απλά βήματα. Και θα το ξαναπώ, αυτό που ήδη κάναν αρκετοί, οι τεχνολογίες δεν μπορούν να αυξήσουν το χάσμα μεταξύ αυτών που μπορούν και αυτών που δεν μπορούν. Θα πρέπει να καλύπτουν τα κενά οι τεχνολογίες. Οπότε θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να καλύψουμε τελείως το χάσμα όσον αφορά ιδιαίτερα ως κοινωνία τις λιγότερο προνομιούχες ομάδες. Τώρα, τι γίνεται με την Ευρώπη. Έχουμε νομοθεσία, έχουμε ιατρικά μηχανήματα που καλύπτονται από την νομοθεσία αυτή. Υπάρχουν και άλλα που δεν είναι ιατρικά μηχανήματα, δηλαδή εφαρμογές που αφορούν το lifestyle, το στυλ ζωής ή άλλα. Νομίζω ότι εμπίπτουν σε άλλες οδηγίες για τα αλλαγματικά προϊόντα, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό, μάλλον ούτε και αυτό έχει συζητήσει αυτό το θέμα και αυτό είναι άλλο ένα μήνυμα που θα επαναλάβω. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε και που μαθαίνουμε στην πράξη. Αυτό που ξέρουμε και υπόθηκε εδώ είναι ότι υπάρχει πολλή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία ας πούμε, των δεδομένων. Έχουμε μια οδηγία για την προστασία των δεδομένων και με τη βοήθειά σας εδώ στο Κοινοβούλιο και με τις εθνικές κυβερνήσεις. Έχουμε κανονισμούς που θα εφαρμοστούν σε δύο χρόνια και βέβαια είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε τώρα για την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών. Εγώ στη χώρα μου, στην Εστονία, ρώτησα τους ειδικούς για τα δεδομένα τι γίνεται με εμά. Και μου είπαν ότι έχουμε καλή νομοθεσία, για τα δεδομένα στην Εστονία, 13 σελίδες. Τώρα έχουμε 300 σελίδες νομοθεσίας που δεν ξέρουμε πώς θα την εφαρμόσουμε. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι θα μάθουμε καθοδόν και τουλάχιστον αν είμαστε συγκεντρωμένοι δεν θα μας αποτρέψει από τη σωστή χρήση αυτών των εργαλείων στο μέλλον. Αν κάποιο λοιπόν θέλει να αποθηκεύσει τα δεδομένα ή έχει άλλε ερωτήσεις, ε, αυτό ήδη απαντάται α πούμε ως ερώτημα. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα δικαιωμάτων χρηστών που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο ήδη. Τώρα στι χώρε μέλη ήμουν στην υποεπιτροπή επίσης για την υγεία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας και οι πληροφορίες μας λένε ότι οι στόχοι που έχουμε είναι σωστοί σε σχέση με αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, προσανατολισμό των ασθενών σε αυτά τα συστήματα, κινητικότητα, μείωση του κόστου κλπ. κλπ. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν και πολλές χώρες που έχουν υιοθετήσει την κινητή υγεία οι μισές από αυτές έχουν κάποιο γενικό νόμο που σχετίζεται με την ψηφιακή υγεία και υπάρχουν κάποια θέματα με τις αδειοδοτήσεις. Θα μπορούσε πάντως ε, κανείς να πει ότι στο ψηφιακό τομέα όσον αφορά το θέμα της ταυτότητας υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή έχουμε δεδομένα από πολλές πηγές, τουλάχιστον στην Εστονία, Δείξω να ισχύει το ίδιο σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντω ω δραστηριότητα έχουν συντονισμό που ξεκινήσει οι χωρε μέλη. Ε, θέλουμε να έχουμε λίγα συστήματα πιστοποίηση. Ευχόμαστε ένα, όχι 27 πια. Και το κυριότερο πια εδώ είναι να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε του επαγγελματίες τη ε, υγεία, γιατί το θέμα με τα δεδομένα αλλάζει συνεχώ. Θα ακούσατε ήδη ότι πολλέ από αυτέ τι δραστηριότητε αφορούν αυτή την ήπια νομοθεσία, το soft law, οι δραστηριότητε συντονισμού ήδη συμβαίνουν. Έχουμε και το κώδικα διοντολογία, ο οποίο θα εγκριθεί, από ό,τι ξέρω, φέτος και ελπίζουμε από το χρόνο οι επιχειρήσει εθελοντικά να αρχίσουν να εφαρμόζουν το κώδικα αυτό. Ολοκληρώνοντα οι πολίτες καθοδηγούν την κοινωνία. Αν θέλετε λοιπόν να ξέρετε κατά πόσο οι λύσεις ταιριάζουν στους στόχους, θα πρέπει να μάθει από πολίτες. Από την εμπειρία, από τις υπηρεσίες και θα πρέπει να τους ακούσετε για το κατά πόσο θέλουν αυτές τις υπηρεσίες. Υπήρξε ένα ερώτημα για το κατά πόσο αισθάνεται άνετα ο κόσμος με την χρήση των δεδομένων. Να σας πω ότι 85% στην Εστονία που ρωτήθηκαν για τις ε, βάσει δεδομένων με στοιχεία υγείας και τα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους έρευνας σε ανώνυμη βάση. Μας είπαν ότι ναι, δεν έχουν αντίρρηση. Παρόμοιε ανταποκρίσει είχαμε και σε άλλες χώρες. Η καινοτομία λοιπόν προέρχεται από τη δράση. Επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά έχουμε πλαίσιο, να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε στην πράξη το πλαίσιο το νομικό από μόνο του δεν να μεταφερθεί από χώρα σε χώρα. Στην Εστονία έχουμε μια νομοθεσία η οποία ταιριάζει με την τεχνολογία και τα πρότυπα διακυβέρνησης που μας επιτρέπουν να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Σε άλλες χώρες όμως το πλαίσιο το νομικό μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες για την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων. Αν ο στόχος λοιπόν είναι σωστός, δεν υπάρχει μόνο μία νομοθεσία, αλλά ένα συνδυασμό νομοθεσία, τεχνολογία και διακυβέρνηση. Και καταλήγοντα να σα πω. Εδώ κάτι που είπε ο Αϊνστάιν. Τα πράγματα πρέπει να όσο πιο απλά γίνεται, αλλά όχι απλούστερα. Να έχουμε ένα στόχο λοιπόν και ένα συμπεφωνημένο και να προσαρμοστούμε. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζει και η συμπεριφορά και η δράση ακριβώς αφορά αυτό το στοιχείο. Να δούμε κατά πόσο δηλαδή ένα πλαίσιο ταιριάζει ακριβώς στους στόχους μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όπως είπατε και στο τέλος της παρουσίασής σας, όταν ε, μελετούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζονται, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στα νομικά πλαίσια, αλλά να μελετούμε το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα νομικά πλαίσια, τις δραστηριότητες των πολιτών, την καλή διακυβέρνηση και στην περίπτωση της Εστονίας είναι πολύ πιο εύκολο γιατί η Εστονία έχει ξεκινήσει το δρόμο της προς το ψηφιακό κόσμο, ε, την πορεία της μάλλον προς το ψηφιακό κόσμο, πολύ πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ψηφιακή, η Ευρώπη πρέπει να γίνει η Εστονία. Είναι πολύ καλό λοιπόν αυτό που έχετε κάνει και βεβαίως είναι πολύ καλό σημείο για τη συζήτησή μας. Για να μάθουμε τι είναι δυνατό να γίνει και ποιοι είναι οι κανόνες που χρειάζονται για να προχωρήσουμε. Επίσης, για να έχουμε πιο ε, ψηφιακά προηγμένες Κοινωνίε. Γιατί όταν μιλούμε για την ηλεκτρονική υγεία, στο μέλλον θα χρειαστεί πιο ψηφιακά προηγμένες κοινωνίες. Χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί. Με ίση πρόσβαση δηλαδή. Για όλους. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στον Μάικλ Παστόρε για τα θέματα αξιοπιστίας. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω με δύο λόγια για την ψηφιακή Ευρώπη. Η ψηφιακή Ευρώπη είναι η φωνή της ε, βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας που εκπροσωπεί περίπου 37 ε, εθνικές ενώσεις και 61 ε, εταιρικά μέρη. Από την αρχή έχουμε εμπλακεί στις δραστηριότητες για την κινητή υγεία, ορίζοντας ποια είναι τα προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί από τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ε, για την ε, πράσινη βίβλο, για την κινητή υγεία που χρονολογείται από το 2014. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα λοιπόν. Η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη των ε, δεδομένων και χρήση τους. Εμπιστοσύνη για την αξιοπιστία των δεδομένων και των... που οσυλλέγουν οι εφαρμογές αυτές θα επικεντρωθώ σε αυτά τα δύο και ευχαρίστω να απαντήσω και σε ερωτήματα για τον κώδικα διοντολογία που εκπονήσαμε και που άκουσα ότι μέχρι το τέλο του χρόνου υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να εγκριθεί. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Θα το δούμε όμω. Τώρα, για την αξιοπιστία των εφαρμογών και τις κατευθυντήρες γραμμές που αναφέρω ο Επίτροπος. Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξουν κατευθυντήρες γραμμές για την αξιοποιηστία των εφαρμογών για αυτά τα δεδομένα που θα τροφοδοτούνται ε, στα ηλεκτρονικά μητρώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, δημιούργησε το μηχανισμό που θα καταλήξει σε αυτές τις ε, κατευθυντήρες γραμμές και φέτος το Μάρτιο η Κομισιόν δημιούργησε μια ε, ομάδα εργασίας ε, εμπειρογνωμόνων ε, που θα εκπονήσει αυτούς τους, αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές και η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της βιομηχανίας όπως εκπρόσωποι της Digital Europe, GSMA και άλλους της κοινωνίας των πολιτών, ομάδων αυτής, ενώσεις ιατρών, ασθενών και περιφερειακούς φορείς, διοικητικούς φορείς, εθνικούς φορείς. Γιατί, γιατί σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρόμοιες δραστηριότητες, οπότε προσπαθούμε να συλλέξουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις συνδυάσουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα μπορεί να ισχύει πανευρωπαϊκά. Ο σκοπός λοιπόν αυτών των κατευθυντηριών γραμμών είναι να μπορούν να τις χρησιμοποιούν οι developers. Δεν είναι βεβαίως υποχρεωτικές. Το Μάρτιο λοιπόν ξεκινήσαμε το εγχείρημα αυτό και ο τρόπος που οργανώσαμε τη δουλειά μας ήταν με τρεις ομάδες. Μία που ασχολήθηκε με το πεδίο εφαρμογή των κατευθυντηρίων, μία που ασχολήθηκε με, το, με τις ομάδες στόχου, ασθενείς, developers κλπ. Και η τρίτη που ασχολήθηκε με τη μεθοδολογία. Πώ θα λειτουργήσουν δηλαδή αυτέ οι κατευθυντήρε γραμμέ από τη δική μα την οπτική, από την οπτική της Digital Europe, αυτές οι κατευθυντήρε θα πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο βασικέ πτυχέ. Η πρώτη είναι το όφελο των ε, δημοσίων αρχών, για να, να αξιολογήσουν δηλαδή την επιστημονική αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγουν αυτές οι εφαρμογές. Η δεύτερη, πιο πρακτική πτυχή, είναι να αποτελέσουν όντως κατεύθυνση, καθοδήγηση έτσι ώστε να ενσωματωθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που συλλέγουν αυτές οι ε, εφαρμογέ και το software που προτείνουν είναι πραγματικά αξιόπιστο. Οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν αρκετές κάποιες αντεφετικές απόψεις, αλλά συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα. Γιατί, Γιατί μιλούμε για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών στην αξιολόγηση κινδύνου και αξιολόγηση συμμόρφωση. Κατά τη δική μα άποψη, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι διαφορέ μεταξύ του τι σημαίνει αξιολόγηση ε, συμμόρφωση που ήδη επιβάλλεται από την οδηγία για, τους, για τις ιατρικές και τον μελλοντικό κανονισμό και την αξιολόγηση Τη αξιοπιστία αυτών των δεδομένων, για την οποία όμως δεν υπάρχει ε, ασφαλέ νομικό πλαίσιο, κάτι που προσπαθούμε να καλύψουμε μέσω αυτών των κατευθυντηριογραμμών. Στην περίπτωση του κώδικα διοντολογία, ε, ε, και στη δική μα την περίπτωση υπήρξαν κάποιες φαίες ζώνες. Είναι δύσκολο να ορίσει κανεί τι είναι η ιατρική συσκευή και τι δεν είναι η ιατρική συσκευή. Βεβαίω. Στι προθέσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής αλλά και τη βιομηχανία και τη Κοινωνία των πολιτών είναι να ξεκαθαριστεί αυτό ακριβώς το κομμάτι. Τι σημαίνει ε, ιατρική συσκευή. Βεβαίως πιστεύουμε ότι το να γίνει η αξιολόγηση συμμόρφωσης ή η αξιολόγηση κινδύνου και να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα σε μια εφαρμογή, κάτι όμως που δεν θα εμπίπτει ε, στον ιατρικό κώδικα δοντολογίας, ίσως να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους ε, developers. Οι μεγάλες εταιρείε έχουν τη νομική δύναμη να, να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, αλλά οι μικροί developers δεν το έχουν. Αυτέ οι κατευθυντήρε γραμμέ λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο σαφεί και απλέ για αυτού για να, τους, να μπορούν να του βοηθήσουν. να κάνω και κάποια σχόλια ακόμη. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι οι κατευθυντές γραμμές θα πρέπει να παραμείνουν, ε, να έχουν στόχο την ε, αποδοτικότητα αυτών των εφαρμογών. Θα πρέπει να συμπληρώνουν την, την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία την οδηγία για τις ιατρικές συσκευέ και να αποτελούν καθοδήγηση για την ε, οδηγία αυτή. Ας πούμε το 2016 για το software. Αν τώρα δούμε την, ε, την διαδικασία συμμόρφωση στα πλαίσια του κατευθυντηρίων γραμμών, μπορεί να δημιουργήσουμε ε, υπερβολικέ απαιτήσει ε, πιστοποίηση. Όπω είπα, υπάρχουν τέτοια εγχειρήματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, εξαιρετικό παράδειγμα στην Ανταλουσία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Έχουμε αρκετά καλά παραδείγματα κατευθυντηρίων γραμμών αξιολόγηση συμμόρφωση για τι εφαρμογέ κινητή υγεία. Αυτέ λοιπόν οι κατευθυντηρίε θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να συμπληρώσουν αυτό που ήδη υπάρχει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ω νομικό κείμενο. Οδηγία, όπω είπα, για τι ε, ιατρικέ συσκευέ και σχετικέ κατευθυντήρε γραμμέ. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσουμε να ζητούμε υπερβολικέ πιστοποιήσει, ε, κινδυνεύουμε να μπερδέψουμε, να συγχύσουμε του ε, developers που θα φτιάξουν τι εφαρμογέ όταν, ε, όταν πρέπει να εντάξουν στο σχεδιασμό του όλε αυτέ τι παραμέτρου. Οπότε θα σταματήσω, Πρόεδρε, εδώ προς το παρόν και αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσω, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα ενδιαφέρει πολλούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Στην αρχή της θητείας, φθινόπωρο του 2014, είχαμε αρχίσει κάποιες συζητήσεις και είχαμε ερωτήσεις και ερωτήματα πρόκυψαν σε σχέση με την ανάγκη τη ρυθμιστική δηλαδή υπήρχε η ιδέα του να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο για ένα κώδικα διοντολογίας να έχουμε μια ήπια νομοθεσία κανόνες αλλά όχι τρακόντια νομοθεσία για να δούμε ακριβώς πώς θα εκλεχθούν τα πράγματα. Και ο Μάρκελ ήταν ε, ακριβώς ένα από αυτά τα άτομα που βοήθησε στο να εμπλέξουμε όλους τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με την Κομισιόν. Θαυμάσιο ήταν αυτό, αλλά βέβαια τώρα πρέπει να θέσουμε νέα ερωτήματα, όπως είπες και εσύ. Κατά τη διάρκεια της εισηγησής σου από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Μήπως έχουν να σχολιάσουν. Γιατί εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι από αυτά τα άτομα που γνωρίζει όλες τις πτυχές του προβλήματος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε σωστή συνεργασία με την Κομισιόν, όταν η Κομισιόν ακριβώς τα γνωρίζει και τα κατανοεί. Η Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Λίγα έχω να προσθέσω σε αυτά που υπόθηκαν στις δύο συνεδρίες. Να σας παραπέμψω στην έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την ηλεκτρονική υγεία και να προσθέσω εδώ μία από τις πέντε συστάσεις που θα βρείτε εκεί για την παιδεία, την παιδεία ηλεκτρονικής υγείας. Και με την εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας. Μαζί με αυτό, να προσθέσω και τη σημασία της ενημέρωσης και οι πολίτες και οι επαγγελματίες της υγείας για τα πλεονεκτήματα και αυτό είναι και όλο το νόημα του ορίζοντα 2020 για την κυκλοφορία αυτών των συστημάτων και την ενημέρωση. Να πω επίσης ότι μέσα στο ορίζοντα 2020 εμείς προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ένωση την Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Το Μάρτι θα έχουμε μία συμφωνία για να συγκροτήσουμε ένα hub στην Ένωση, δουλεύοντα διτά, συλλέγοντας πληροφορίες ιατρικές και αποδεικτικά στοιχεία όπω υπόθηκε στην αρχή και δεύτερον, να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη στην εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Τέλος, να πω ότι όπως είπε και ο κύριος Μπόνι ανακύπτουν νέα πράγματα μέσω συζήτησης, μέσω εξέλιξης και η κινητή υγεία είναι, ένα, είναι τμήμα της, του σχεδίου δράσης που εθετήσαμε το 12. Σχέδιο δράσης που αφορά την περίοδο 12 με 20. Θα κάνουμε μια διάμεση αξιολόγηση και στο τέλος του έτους μέσω διαβούλευσης θα ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι νέοι τομείς όπου θα πρέπει να έχουμε περισσότερες γνώσεις ή ποιοι είναι οι τομείς με τους οποίους δεν ασχοληθήκαμε καθόλου μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και ο Πρόεδρος. Έχουμε τον κύριο Κόβλητσε και, το, και την κυρία Βέρνη, ευρωβουλευτές. Αν θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς ή αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, είτε να πείτε και τις απόψης σας. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ρωτήσω το θέμα που συζήτησε ο κύριος Αβιξόν από την Εστόνια, ποια είναι τα επόμενα βήματα του ενοποιημένου πρωτοκόλλου, γιατί αυτό θα αποτελέσει ένα από τα θεμέλια του όλου πράγματος για να συλλέξουμε δεδομένα και να τα χρησιμοποιούμε από απόσταση θα πρέπει να ε, βασίζονται αυτά σε ένα ενοποιημένο πρωτόκολλο. Γιατί αλλιώς τα μηχανηματάκια δεν θα λειτουργούν, δεν θα συνεργάζονται μεταξύ τους Θα το γνωρίζετε αυτό στην Εστονία καλύτερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι έχετε πλήρη ηλεκτρονική διοίκηση. Έχουμε προβλήματα παρόμοια εμείς στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία, το βασικό πρωτόκολλο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στα αγγλικά ή αν θα κωδικοποιούνται δεδομένα με κάποιο τρόπο, αν θα κωδικοποιούνται στα λατινικά, με ενοποιημένη ορολογία, γιατί ούτω ή άλλω οι γιατροί ανά πάσα στιγμή μπορούν να συζητήσουν μεταξύ του χρησιμοποιώντα τη λατινική. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα, από το οποίο θα εξαρτηθούν όλα τα υπόλοιπα. Χρειαζόμαστε ένα ενοποιημένο πρωτόκολλο που να λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αβέρνη. Μήπως έχετε να προσθέσετε ή να ρωτήσετε κάτι. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε στην Ευρώπη των 28. Μιλάμε διάφορες γλώσσες και στις εφαρμογές και παντού στο σύστημα θέλουμε να χρησιμοποιηθεί σε όλε τι χώρε. Αλλά ο κόσμο έχει τη δικιά του γλώσσα. Ε, έχουμε ακόμα θέματα υγείας. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε και μεταφράσουμε αυτά τα εργαλεία στις διαφορέ χώρε. Ευχαριστώ. Αν συμφωνείτε, έχουμε χρόνο για ανοιχτή συζήτηση. Ας ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Το κοινό μπορεί να θέσει ερωτήματα, λέει ο Πρόεδρος. Απευθύνομαι σε όλους σας, έτσι. Όλους τους παρόντες στην αίθουσα. Πείτε μας αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια. Παρακαλώ. Θα σας ζητήσω να μας συστηθείτε πρώτα. αυτό λέτε, από τη Γερμανία. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι σημαντικό και που αφορά την Εστονία, την οποία ζηλεύουμε εμείς στην Γερμανία για αυτά που έχουν κάνει. Το βιβλίο σας ονομάζεται «Πανασχεδιάστο τέλο πάντων την παροχή υγείας στην Ευρώπη με ως 2020». Κάτι τέτοιο είπατε. Ναι, πραγματικά πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα συστήματα υγείας. Και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών αλλάζει και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αφορά επίσης το στοιχείο της εκπαίδευσης στην υγεία, ασφάλειας, υγείας, οργάνωση των νοσοκομείων, όπου δεν έχουμε κοινό πεδίο. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο η Κομισιόν του το Κοινοβούλιο εδώ θα μπορούσαν να έχουν περισσότερο καθοδηγητικό ρόλο. Η απάντηση που ακούμε είναι συνέχεια βέλτιστες πρακτικές. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι στο τομέα της υγείας βέλτιστες πρακτικές σημαίνει ότι έχουμε τελείως διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούνται. Και το πράγμα της Ιστονίας δεν μπορεί ας πούμε, να το πάρουμε copy-paste στην Γερμανία για διάφορους λόγους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μήπως κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Ο συνάδελφος από την Κομισιόν. Ναι. για αυτές τις ορολογίες. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα το λέμε στη δικιά μας αργό. Αναφέρθηκαν τα λατινικά ως lingua franca της ιατρικής επιστήμης. Στην ιατρική όμως υπάρχουν πολλοί τρόποι να διασφαλίσουμε ότι μιλάμε για τα ίδια Βεβαίω υπάρχει και η διεθνή ταξινόμηση ασθενειών που μα διευκολύνει. Τώρα αυτό που αναπτύσσουμε είναι πολύ πιο περίπλοκο ως λεξιλόγιο. Έχουμε μια κλινική ορολογία που καλύπτει 500.000 έννοιες και τις σχέσεις τους και είναι τελείως ψηφιοποιημένο. Πάω στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν εφαρμόζουμε ακόμα αυτή την ορολογία, αυτή τη νόμη, όσο και αν ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Αυτά που ανέφερε προηγουμένω ο Επίτροπο, την ηλεκτρονική δηλαδή μετάδοση διασυνοριακά των συνταγών και των φακέλων και τα δύο δίνουν έμφαση σε αυτό το πρόβλημα και το πώς ακριβώς ας πούμε μπορούν οι συνταγές, οι συνταγογραφήσει να μεταφερθούν από χώρα σε χώρα. Αυτό ξεπερνάει τη σημασιολογία και θεωρούμε ότι εύκολα μπορεί να λυθεί. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε τοπικά αλλά όχι παγκοσμίω. Και πρέπει να ρυθμίσουμε αυτά τα δύο σε αυτή τη φάση. Βέβαια υπάρχουν όμως και άλλες εξελίξεις. επιστήμη των υπολογιστών, η οποία μας βοηθάει. Και οι αυτόματες μεταφράσεις. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της μασοξιολογικής λειτουργικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα χρόνο για άλλες ερωτήσεις αν θέλετε. Παρακαλώ. Γεια σας. Από τις Βρυξέλλες στο Μακεδονά. Ένα σχόλιο περισσότερο παρά ερώτημα. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση για την κινητή υγεία. Ο κύριος Κασιανός και ο κύριος Παστόρε στις εισηγήσεις τους, ακούγοντάς τες, είχα την εντύπωση ότι αυτό το θέμα είναι πολύ λεπτό, γιατί αφενός χρειαζόμαστε να μιλήσουμε κάτι το οποίο ρυθμίζεται πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφενός και αφετέρου υπάρχει το ερώτημα ή το ζήτημα της βελτίωσης της καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ακούσω λοιπόν από εσά σε σχέση με την μελλοντική ανάπτυξη αυτών των εργαλείων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο τώρα οι υπόλοιποι. Το κοινό. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ωραία. Επανερχόμαστε σε εμά λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα οι εισηγητές μα να σχολιάσουν αυτές τις ερωτήσει ή τις παρατηρήσεις που ακούσαμε και να αναπτύξουν κάποια άλλα θέματα αν θέλουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, uh, Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τα βανή από πλευρά Κομισιόν που αρχίζετε να εισάγετε αυτό το θέμα το ερώτημα του πώς οι διάφορες, ε, άνθρωποι από διάφορες χώρες με διάφορες γλώσσες θα κατανοήσουν ένα στον άλλο θα γίνεται κατά περίπτωση. Δεν θα υπάρχει πρώτα κάποιο είδους ε, κοινό ενοποιημένο πρωτόκολλο, αλλά μια διαδικασία όπου υπηρεσία κατά υπηρεσία θα μπορούσαμε το, θα αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο, ας το ονομάσουμε έτσι. Κάποιες ε, κατατάξεις είναι παγκόσμιες κατατάξεις ασθενειών αλλά για να γίνει και τόσο απλό όσο μια συνταγογράφηση κατανοητή στη Φιλανδία στην Ελλάδα θα πρέπει να αναπτυχθεί, να πλήρως. Οπότε αυτό ακριβώς θα γίνει. Οι χώρες έχουν συμφωνήσει πολλές από αυτές να εγκαταστηρίσουν αυτή την διασυνοριακή υπηρεσία. Το 2018 έχει δώσει κονδύλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό, οπότε πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικότητα γιατί τόνισα τόσο πολύ τη συνιστόσα του ασθενούς. Και αναφέρθηκε κιόλα ότι η μεταμόρφωση του συστήματος υγειονομική περίθαλψης είναι κάτι σημαντικό. Η δύναμη προέρχεται από δύο βασικές πηγές, το χρήμα και τις πληροφορίες. Για να ενδυναμώσουμε λοιπόν τους πολίτες, να τους χειραφετήσουμε, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε τη χειραφέτηση από τους επαγγελματίες της υγείας. Απλά να την κατανέμουμε ισότιμα στους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία που βασίζεται σε αυτά τα χρήματα και τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθάλψης και γνωρίζω από πολλούς φίλους και συναδέλφους ότι φοβούνται ότι οι ασθενείς δεν θα καταλαβαίνουν και θα υπάρχει αυξημένο κίνδυνο συνεπώ του τι θα γίνει αν μάθουν περισσότερα για την υγεία τους. Αυτό έχει ήδη δοκιμαστεί. Ο κόσμος δεν βλέπει ως αποτρεπτικό ούτε καν τον επιπλέον φόρτο εργασία εφόσον υπάρξει ευαισθητοποίηση ταυτόχρονα. Και ευχαριστώ που το αναφέρατε αυτό. Είναι ακριβώς αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κομισιών αλλά και στα κράτη-μέλη. Μετά ε, ε, άκουσα μια ερώτηση για την παρουσίασή μου κατά πόσο ε, μπορεί να επιτελέσει τους σκοπούς. Εάν συμφωνήσουμε επί ενός σκοπού, δηλαδή τον επανασχεδιασμό των συστημάτων υγειονομικής περιθάλψης, ε, με ανάγκη χειραφέτηση των ασθενών, τότε δεν χρειάζεται να ξαναθέσουμε το ερώτημα του αν υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα στην χρήση των ασθενών. Έχουμε ένα κανονισμό που λέει ότι πρέπει να κάνει κάποιο ε, επιλογέ βάση ενημερωμένε και έχουμε την εμπειρία από την Εστονία και από άλλε χώρε για το πώ πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Στην Εστονία ένα τρόπο είναι να είναι όλα διαφανείς. Στη δική μα πύλη για την υγεία όλοι οι ασθενεί μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του. Προς το παρόν σκοπός είναι η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, γράφει κάτι ο οικογενειακός γιατρός για τον ασθενή και μετά ο ειδικό, ο ειδικευμένος γιατρός ε, μπορεί να δει αυτές τις πληροφορίες και το γνωρίζει ο, ο ασθενής ότι έγινε τέτοια γνωστοποίηση πληροφοριών και μπορεί να γνωρίζει ο ασθενή όταν τα δεδομένα του χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικού σκοπού. Αν να διδάξουμε λοιπόν του ασθενεί ότι όλο αυτό γίνεται προ όφελό του και ότι μπορούν μέσω τη έρευνα να συμβάλλουν για το καλό των υπολείπων, τότε το όραμα του Επιτρόπου Ανδριουκάητη ε, για ε, ε, ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων το οποίο θα μπορεί να κοινοποιηθεί σε πολλέ χώρε. Και ξέρω ότι η Δανία και η Φιλανδία έχουν συμφωνήσει να φτιάξουν κάτι μεταξύ του. Η Εστονία πραγματεύεται επίσης με τις σκανδιναβικές χώρες. Είναι λοιπόν κάτι δυνατόν, αλλά μόνο εάν είμαστε βέβαιοι ότι ο κόσμος το επιθυμεί και αν γίνουν κάτι παρόμοιο αργότερα, δηλαδή ότι συνεχώς θα παρακολουθούμε το όλο νομικό πλαίσιο και το πώς εφαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο και να υπάρχει και δυνατότητα να κάνουμε αλλαγέ ξεκινώντα με την ήπια νομοθεσία, εφόσον θεωρήσουμε ότι υπάρχει λόγος ε, να αναλάβουμε πιο αυστηρή ε, πιο δράση. Τότε μπορούμε. Ε, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε να υπάρχουν εμπόδια για να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Ναι, Μικέλα. Έχω μερικά σχόλια όσον αφορά το ζήτημα της κινητής υγείας και της ρύθμισής της ή της υπερβολικής της ρύθμισης. Ναι, Πραγματι είναι ένα τομέα που ρυθμίζεται υπερβολικά και αυτό είναι καλό. Ένα παράδειγμα, όσον αφορά τα ε, στοιχεία, τα δεδομένα και την κοινοποίησή τους. Επειδή το αναφέρατε, όσοι ε, γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία, τα δεδομένα ρυθμίζονται πολύ αυστηρά. και σε εθνικό επίπεδο με διάφορες διατάξεις ε, οι οποίες ποικίλουν από κράτος σε κράτος. Ένα πράγμα που εμείς ε, διαρκώς υποστηρίζουμε είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε μια δεσταυρούμενη ροή δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα δεδομένα υγείας. Αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα ως δομή που θα υποστηρίζει μια ένα πανευρωπαϊκό σύστημα υγείας. Εμείς ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα εμπιστοσύνη στον κώδικα δεοντολογία που ανέφερα. Προσπαθούμε δηλαδή στον κώδικα δεοντολογία να συμπεριλάβουμε στοιχεία τα οποία θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών αλλά και θα βοηθήσουν του προγραμματιστέ να προγραμματίσουν τι σωστέ εφαρμογέ συλλογή ε, δεδομένων υγεία των χρηστών. Όσοι από εσά δεν το έχετε δει, σα συνιστώ να ρίξετε μια ματιά, διότι εμεί πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα βήμα προς τα εμπρό σε σχέση με άλλε πρωτοβουλίες. Όσον αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων, όπως αναφέραμε στη συζήτηση εδώ στο πάνελ, τα δεδομένα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να είναι αξιόπιστα. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε και θέλουμε να προτείνουμε θα είναι ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών. Πώ δηλαδή σε εθνικό επίπεδο αλλά και πώ οι επιχειρήσει προσπαθούν να επιτύχουν αυτή την επιστημονική εγκυρότητα των δεδομένων. Όλα δίνα, σύμφωνα με του υπάρχοντες κανονισμού. Και πάλι ήθελα να επισημάνω ότι ο hard law τόσο από την άψη των δεδομένων ε, υγείας όσο και από την άψη της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για ιατρικές εφαρμογές ή όχι. Αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία μια εφαρμογή συλλέγει αυτό που εμείς βλέπουμε ή που καθορίζουμε ως δεδομένα για να οριστεί μια εφαρμογή ως ιατρική. Τα δεδομένα που συλλέγει μια εφαρμογή δεν καθορίζουν τη φύση μιας εφαρμογής ε, ως ιατρική ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για την αξιοπιστία, για την ε, επιστημονική εγκυρότητα των δεδομένων αυτών. Γι' αυτό το λόγο ε, διασταυρώνονται αυτές οι δύο πτυχές και είναι διασυνοριακές. Ευχαριστώ. So I think that now we will... Ωραία. Ας προσπαθήσουμε τώρα να συνοψίσουμε τη συζήτηση. Ε, έχετε το λόγο ε, εκ μέρους της ΕΜΒΗ και της... Ε, Ευχαριστώ, Μιχάλ. Δεν είμαι πολύ καλός στα λατινικά, αλλά μπορώ να πω στον κύριο Καοχλιτσέκ ότι η lingua λατίνα πουλχρα έστ. Είναι μια πρόκληση να, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο του να αντικαταστήσουμε λόγω του Brexit την Αγγλική με τη Λεθνική. Να μην μπω σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, το πιο ευχαριστώ μέρο τη ημέρα ήταν αυτέ οι δύο ώρε που πέρασα εδώ και ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Με τις τρεις μου ιδιότητες. Ως πολίτης, ε, χαίρομαι με την προοπτική της κινητής υγείας όπως παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εδώ. Έμαθα πολλά πράγματα εδώ που θα με βοηθήσουν ε, να ενημερωθώ, να αξιολογήσω και ελπίζω ότι στο μέλλον θα σπαταλώ λιγότερο χρόνο και λιγότερο χρήμα για την υγεία μου. Και θυμάμαι πριν κάποιε δεκαετίε, όταν η μητέρα μου ή ο πατέρα μου έπρεπε να πάνε να ελέγξουν την πίεσή του, χρειάζονταν μια ολόκληρη ημέρα. Γιατί εμεί ζούσαμε σε ένα χωριό και χρειαζόμασταν δύο ώρε με τα πόδια για την κοντινότερη πόλη. Και τώρα ε, παίρνει κανεί την πίεση του σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πρόκειται για επανάσταση. Και είμαι και ευγνώμων ε, ως μέλος ενός ε, εδώ ενό νομοθετικού σώματο που μαθαίνω περισσότερα. Πολλά πράγματα υπάρχουν εδώ να μάθουμε. Και μερικές φορές η εξέλιξη ξέρετε, είναι ταχύτερε από τους νομοθέτε. Οπότε ευχαριστούμε που μας διαφωτίσατε, μας κάνετε μια τόσο καλή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Ήθελα να πω ότι πολλοί δομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας ικανοποιούν όσον αφορά τα αποτελέσματα που παρέχουμε. Αλλά εδώ στον τομέα της υγείας, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερη αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν νομοθετούμε, τα πράγματα λειτουργούν. Και το ψηφιακό θεματολόγιο είναι ένα από αυτά. Και αυτό που χρειάζεται πιστεύω είναι να συνεχίσουμε ε, να παρέχουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ενδεχομένως να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι στην ερμηνεία της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την υγεία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Και οι πολίτες ε, αναμένουν να κερδίσουν και κάτι από το γεγονός ότι 28 χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα πρέπει αυτό να προσθέσει αξία στη ζωή τους. Εδώ πιστεύω λοιπόν ότι μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη προστάμινη αξία. Αισθάνομαι πιο αισιόδοξο μετά από αυτή τη ε, συνάντηση εδώ. Και θα ήθελα να κλείσω παραθέτοντας τα λόγια του Επιτρόπου που είπε «Έχει έρθει η ώρα, ας αξιοποιήσουμε τη στιγμή, την ορμή που έχουμε αυτή τη στιγμή». και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από πλευράς ΕΝΒΙ για όλες τις συμμετοχές και για την παρουσία όλων σας και ειδικότερα θα χρησιμοποιήσω τη σλοβενική μου πλευρά να καλωσορίσω μια ομάδα νέων Ευρωπαίων από τη Σλοβενία που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω ότι η MVK οργανώσαμε μία εξαιρετική ακρόαση η οποία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ήθελα να μοιραστώ με σας μερικές σκέψεις ε, εν είδη συμπερασμάτων από την ανταλλαγή απόψεων σήμερα και από τις συζητήσεις μας. Πρώτα απ' όλα, Όλοι αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω, ότι ζούμε σε εποχές όπου τα συστήματα υγείας αλλάζουν. Πρόκειται για μια μετάβαση από ένα παραδοσιακό μοντέλο υγειονομικών συστημάτων που αντιδρούσαν σε κάθε ασθένεια, σε ένα μοντέλο όπου η οργάνωση των ε, συστημάτων υγείας ε, επικεντρώνεται περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για την ποιότητα ζωής. Δεύτερον, συζητήσαμε πολλά θέματα που αφορούν ιατρικά μηχανήματα, εφαρμογές ε, και εφαρμογές που δεν είναι ιατρικά μηχανήματα που ε, ε, ε, επιδελούν απλά ψυχαγωγικό σκοπό. Αλλά ξέρετε, αυτές οι εφαρμογές σχετίζονται με το ιατρική. Συχνά δημιουργούν νέες στάσεις, νέες, νέα ανάληψη ευθυνών από εμάς τους ίδιους πολίτες, ως χρήστες, ως δυνητικοί ασθενείς. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να ε, εντοπίσουμε ποιο κομμάτι αυτών των ε, λύσεων ε, που χαρακτηρίζουν αυτή τη μετάβαση πρέπει να ρυθμίζονται αυστηρά με αυστηρούς κανόνες και ποιο κομμάτι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κάποιους κοινούς κανόνες θα χαρακτηρίζονται από έναν κώδικα διοντολογία, κατευθυντήρε γραμμέ, αυτορύθμιση. Διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε κατά τη συζήτηση. Δεν πρέπει να σκοτώσουμε την καινοτομία, αλλά να την υποστηρίξουμε. Τρίτον, εδώ μιλάμε για ιατρική βασισμένη καθοδηγούμενη από τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που θα γίνει με τα δικά μας στοιχεία, τα στοιχεία υγείας μας ε, και άλλα προσωπικά δεδομένα. Ε, τα δεδομένα των πληθυσμών, ε, των λαών και Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, τον κανονισμό γενικής προστασίας των δεδομένων, την ανωνυμοποίηση, την ψευδονυμοποίηση. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι από τη μια πλευρά έχουμε την προστασία των ατομικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη μας ως ασθενείς, αλλά και από την άλλη έχουμε την ασφάλεια των συστημάτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων ταυτόχρονα για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Προηγουμένως ε, αναφέρθηκε ότι χρειαζόμαστε κάποιο είδους παιδεία για την ψηφιακή υγεία. Πιστεύω ότι αυτή η παιδεία για την ψηφιακή υγεία είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους γιατρούς. Για όλους μας. διότι πρέπει να συνομιλούμε σε μια κοινή γλώσσα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο και τα προβλήματά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα καθηκοντά μας που θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας απασχολήσει, να το σκεφτούμε πώς θα αναπτύξουμε αυτή την παιδεία για την ψηφιακή υγεία γιατί θα αποτελέσει θεμέλιο για αξιόπιστες λύσεις ε, πανευρωπαϊκές. Πέμπτον, χρειαζόμαστε κάποιες προϋποθέσεις και το είπαμε όλοι οι υποδομές είναι αδύνατον να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες που θα αντιδρούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου χωρίς την τεχνολογία 5G με το πάρα πολύ γρήγορο διαδίκτυο στο μέλλον. Και δεν μιλάμε για το 2050, μιλάμε για τα χρόνια που έρχονται τώρα. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και από την άλλη διαλειτουργικότητα. Υψηλό επίπεδο με αυτές τις σημειολογικές ε, λύσεις που μας θα δώσουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε και να μεταφράζουμε τις πληροφορίες. Στην Ευρώπη Εργαζόμαστε για τη διαλειτουργικότητα, υποστηρίζουμε κάποια προγράμματα και κάποιες διαδικασίες και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν. Εναρμόνιση των κανόνων επίσης κανόνας τα ε, η, προστασία των... η γενική προστασία των δεδομένων, αλλά όχι μόνο. Ε, ξέρουμε όλοι μας ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πανευρωπαϊκά θα είναι δυνατή εφόσον πληρείται αυτή η προϋπόθεση. Το ίδιο ισχύει για την πιστοποίηση, για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και για τη συνεργασία των ενδιαφερομένων ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές και κοινωνικές προϋποθέσεις ε, για ε, ό,τι θα γίνει στο μέλλον. Έκτον, κάποιος το υποστήριξε στεναρά για να επιτύχουμε τους στόχους μας και να αποτελέσουμε υπόδειγμα ε, μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας. Όπως είπε και ο Επίτροπος, αυτές οι κοινέ προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών ε, και σε συνεργασία με την Ελβετία στο ΣΕΡΝ χρειαζόμαστε αυτές τις νέες γνώσεις γιατί αυτές οι νέες γνώσεις θα μας ε, δώσουν νέες δυνατότητες εξατομίκευσης των θεραπείων. Η εξατομίκευση σε αυτό το τομέα δεν ούτε εξατομίκευση σε άλλες υπηρεσίες όπου βέβαια είναι σημαντική, αλλά σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική διότι θα δώσει τη δυνατότητα εξατομικευμένης θεραπείας προσαρμοσμένη στις πραγματικές μας ανάγκες ε, που θα βασίζεται στη σωστή ενημέρωση περί της κατάστασης της υγείας. Έβδομον, όπως ακούσαμε από πολλούς, μετά από όλα αυτά θα πρέπει να φτιάξουμε ένα κατάλογο του τι προγραμματίζουμε να κάνουμε και σε τι χρονοδιάγραμμα. Γίνονται διάφορες προσπάθειες φυσικά από την Κομισιόν και αυτό μας δείχνει τη στρατηγική υπάρχει, Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να καταρτήσουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, μια νέα ατζέντα για τι μελλοντικέ μα δραστηριότητε και ορισμένα που μα θα πρέπει να επιταχύνουμε τι προσπαθίε μα. Όγδον, ήθελα να πω πόσο καταπληκτικό είναι που ε, ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου από την Ήτρε και την Έμβη συνευρίσκονται εδώ είναι σημαντικό γιατί μας δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε την ολιστική διάσταση της υγειονομικής περίθαλψης για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία σκεπτόμενη δημόσια πολιτική και ασθενείς. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το δεχόμενο κάποια εκθέσει πρωτοβουλία που να αφορά αυτέ τι δραστηριότητε που προετοιμάζει η Κομισιόν. Ένατον. Ορισμένοι υποστήριξαν στεναρά ότι πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και ότι θα πρέπει να προσέξουμε ε, τι γίνεται όσον αφορά τις τιμές. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν την ευαισθητοποίηση, τιμές προσιτές σε όλους και προσβασιμότητα για να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ. Ήταν ε, πολύ ευχαριστή η παρουσία σας εδώ και πολύ χρήσιμη που συζητήσαμε αυτή την νομοδότηση. Ε, μας δόθηκε η ευκαιρία να κοιτάξουμε κάποιες ιδέες ε, όπως τις βλέπουμε από την οπτική γωνία του κράτους όταν ε, συνδυάζουμε τις κρατικές δραστηριότητες με τις νέες τεχνολογικές λύσεις από την οπτική γωνία των επιχειρήσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την οπτική γωνία των ερευνητών για να κατανοήσουμε και τις προκλήσεις, τι δημογραφικές προκλήσεις ε, και πώς αυτή η νέα μεταμόρφωση της υγείας θα, χρησιμοποιήσει, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την γύρανση του πληθυσμού μας με προληπτικές λύσεις, πιο προληπτικές, αλλά και πρακτικά με αυτή την ε, πρόταση μιας πλατφόρμας τηλεϊατρικής για πρακτική χρήση. Όλες αυτές οι πτυχές λοιπόν, όλες αυτές οι διαστάσεις πιστεύω είναι σημαντικές και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους, την Ήτρε, την Έμβη, όλους τους συναδέλφους μας και σας παροτρύνω να συνεχίσουμε αυτό το έργο μαζί, όλοι μαζί, ως κοινή ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ.